Okay, can we try... Εντάξει λοιπόν. <laughs> Για να δοκιμάσουμε λέει ο Πρόεδρο. Εντάξει, οι καμπίνες διερμηνίας γνέφουν θετικά, άρα είμαστε εντάξει νομίζω. Λοιπόν, ο κύριος Βαντάλαν θα αναλάβει την προεδρία αργότερα, αλλά ας αρχίσουμε πρώτα, πρώτα με την ε, συμφωνία με το Βιετνάμ Η συμφωνία αυτή με το Βιετνάμ είναι κομμάτι των κλασικών συμφωνιών που αντικαθιστούν τις εθνικές ε, συμφωνίες. Στο Συμβούλιο έγιναν μεγάλες ε, διαπραγματεύσεις και μακρόχρονες διαπραγματεύσεις. Υπήλθε συμφωνία, αλλά δεν ε, επήλθε συμφωνία για τη φορολόγηση των καυσίμων, γιατί δεν συμφώνησε το Βιετνάμ. Ωστόσο τα άλλα θέματα ε, συμφωνήθηκαν θα πρέπει λοιπόν να, συμφων... συζητηθεί αυτό το θέμα με τα κράτη-μέλη. Τώρα, γιατί υπάρχει και μια άλλη δυσκολία με τις Ηνωμένε Πολιτείε σχετικά με τις εναέριες μεταφορές ε, και... Αλλά ε, προτείνεται να ε, υπερψηφιστεί η συμφωνία αυτή εκτός από το κομμάτι που είναι μια στάνταρ συμφωνία εκτός από το κομμάτι για τα καύσιμα. Yeah, Ευχαριστώ πολύ Ντομινίκ, Λέω ο κύριος Βαντάλ. Αρχίζουμε τώρα λοιπόν τους κοιόδης, κυρία Τικάου. Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα σε σχέση με αυτή την έκθεση. Είναι γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα με την φορολόγηση όχι όλων των καυσίμων, αλλά ειδικά της κυροσύνης που χρησιμοποιούν τα αεροπλάνα. Αλλά καταρχήν υποστηρίζουμε την έκθεση Ρίκε και είμαι πεπισμένη ότι και σε για πολλές άλλες συμφωνίες που βρίσκονται στην ε, ημερήσια διάταξη θα μπορέσουμε να δώσουμε το πράσινο φως σήμερα. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Μάισνερ, ε, εκ μέρου των φιλελευθέρων. Ναι, συμφωνώ. Α, βέβαια, καλύτερα θα ήταν να είχε εγκριθεί και το κομμάτι της φορολόγηση των καυσίμων, αλλά όπως είπε και η κυρία Τικάου, σε σχέση με άλλε συμφωνίε είναι α, πολύ καλή τούτη εδώ η συμφωνία. Οπότε, ε, συμφωνούμε. Δεν ξέρω, λέει ο κύριος Βαντάλ. Θα ήθελα να παρακαλέσω Oké, okay, ik krijg een duim omhoog, dus we kunnen verder. Kennelijk werkt alles weer. Dan hebben we nu mevrouw Lichtenberger. Dem Abkommen zu Vietnam kunnen we zustimmen. Μπορούμε να συμφωνήσουμε, λέει η κυρία Λίχτενμπεργκερ, για τη συμφωνία με το Βιετνάμ. Πάλι πρόβλημα, λέει. Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κυρία Λίχτενστάιν. Προχωρούμε. Φόρστερ. Όλα. Άλλε είναι όρντνουγ, λέει η κυρία Φόρστερ. Συμφωνούμε. Θα συμφωνήσουμε με τον εισηγητή. Πολύ ωραία, λέει ο πρόεδρος. Υπάρχει κανείς εδώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα μπορούσε να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Ρίκε για την έκθεσή του. Είναι σημαντική έκθεση αυτή, είναι σημαντικό να εγκριθεί η συμφωνία γιατί ευθυγραμμίζεται το απονομική ε, από νομική άποψη το δίκαιο που ισχύει. 17 ξεχωριστές συμφωνίες υπήρχαν και Βεβαίω δεν είναι 100% παραδοσιακή και στάνταρ η συμφωνία αυτή γιατί δεν έχει τη ρήτρα για τη φορολόγηση των καυσίμων αλλά είναι πολύ καλή. Συμφωνούμε. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ ο εισηγητή για να κλείσει ο κύκλο. δεν έχω τίποτα να συμπληρώσω λέει ο εισηγητή. απλώ να ευχαριστήσω ε, και την Κομισιόν για τη θέση τη και του συναδέλφου. πολύ ωραία πολύ αποτελεσματικός τρόπος αυτός βεβαίως δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε την έκθεση αυτή καθεαυτή, δεν μπορούν να υποβληθούν τέτοιου είδου τροπολογίε αλλά μπορούν να υποβληθούν άλλου είδου τροπολογίε για τη διαδικασία μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου. Στις 28 Φεβρουαρίου πάει το θέμα στην Επιτροπή και ελπίζουμε να προχωρήσει στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Αυτά για τη συμφωνία ε, με το Βιετνάμ ε, για τις αεροπορικές μεταφορές προχωρούμε στην έκθεση του κυρίου Σαζάντα τροποποιητικό πρωτόκολλο της συμφωνίας με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Ο συνάδελφος Ασάντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το πρωτόκολλο το οποίο συζητούμε εδώ είναι ιδιαίτερη σημασίας στις αγορές αναέριων μεταφορών και, των, ε, και της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών και καλύπτει ουσιαστικά το 60% των αεροπορικών μετακινήσεων. Υπάρχουν διατάξεις στο πρωτόκολλο αυτό για τη μη διάκριση και για την παροχή αν θέλετε κάποιων α, ωφελών προς όλους και προς τους αεροπορικές εταιρείες αλλά κυρίως προς τους επιβάτες. Ε, το όνειρό μας είναι να βελτιώσουμε τα πράγματα για τους καταναλωτές, να έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα και να, να η διαδικασία. Βέβαια στο πρωτόκολλο δεν εγγυάται όλο, όλα αυτά αλλά είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε επίσης ε, πλήρως το όλες τις πτυχές που αφορούν τους επιβάτες ε, στη, είχαμε την έκθεση Simpsons για τις βίζες ε, και τα λοιπά στο παρελθόν που συζητούσαμε αυτά είναι όλα συμφαν... συναφή θέματα μπορούσε να φανταστεί κανεί για τις αεροπορικές μεταφορές το, το πρωτόκολλο δεν ασχολείται με τέτοια θέματα αλλά ε, υπάρχει εδώ μια σημαντική ρήτρα Δίτρα Αναστολής η οποία ομοσδιούχοι πολλών εν λόγω αεροπορικών εταιρειών που είναι συνδεδεμένοι η οποία άλλες σημαντικές οι δίτρα Αναστολής μες για ένα χρόνια α, πίσω γιατί Υπάρχει ουσιαστικά αδυναμία πτήσεων από ορισμένε χώρε προ τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, δυστυχώς το πρωτόκολλο αυτό δεν επιλύει τέτοιου είδους θέματα ε, τα θέματα, τα προβλήματα που είχαμε ε, έκλεισαν οι διαπραγματεύσεις οι σχετικές θα μπορούσαμε βεβαίως να χρησιμοποιήσουμε την κοινή επιτροπή η οποία συμφώνως προς το άρθρο 5 ενδεχομένως θα μπορούσε να επηρεάσει τα πράγματα Και βεβαίως η Επιτροπή αυτή θα ίσως θα προσ... μπορούσε να τροποποιήσει περαιτέρω κάποια πράγματα Θα ήθελα τώρα να σχολιάσω ορισμένα πράγματα που είπαν οι σκιώδεις εισηγητές. Ε, συμφώνησα βεβαίως ότι πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά ο κύριος Λάιχφριτ παραδείγματος χάρη ανησυχεί για το ότι ακόμη και στη δεύτερη αυτή φάση δεν ανοίγουν 100% οι αγορές. Είναι αλήθεια αυτό, αλλά ε, ξεκινάνε κάποιες μεταρρυθμίσεις νομίζω ε, και βλέπουμε να υπάρχει δυνατότητα για ευρωπαϊκές εταιρείες να αποκτήσουν μερίδια πλειοψηφιακά στις ε, Ηνωμένε Πολιτείες. Κατά αντιστοιχεία βεβαίως θα πρέπει και οι αμερικανικές εταιρείες να έχουν το δικαίωμα αυτό στην Ευρώπη. Ίσως είναι ανισομερής η κατάσταση ακόμη και οι διαπραγματεύσεις δεν μπόρεσαν να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα αλλά τέλος πάντων θα δούμε τι θα γίνει. Ο κύριος Ελκαντράουι έκανε ορισμένα σχόλια για τα οποία τον ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα εγώ να ε, κάνω μια, ε, να υποβάλω ο ίδιος μια τροφ, πρωτοβουλιακή τροπολογία στην δική μου την έκθεση γιατί η έναρξη μιας νέας φάσης διαπραγματεύσεων σημαίνει ίσως διαφορετικά πράγματα στα πολωνικά από ότι στη, σε άλλες το κατανοούμε αλλιώ αυτό. Χαίρομαι γιατί ε, στην, ε, ε, τώρα εισήχθη στο πρωτόκολλο ένα, μια παράγραφος για τα κοινωνικά θέματα Και βεβαίως Ε, έγιναν και διάφορα σχόλια από τους φιλελεύθερους στους οποίους θα ήθελα να απαντήσω ότι ήδη έκανα κάποιες αλλαγές στο κείμενο και ζητώ πλήρη απελευθέρωση, προστασία για τους επιβάτες κτλ. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να καλύπτει κάποιες ανησυχίες των φιλελεύθερων. Τώρα ερχόμαστε στο ακανθόδες θέμα της ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων με, τους, με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η ανταλλαγή θα πρέπει να γίνεται στην αμοιβαία, με βάση την αμοιβαία αναγνώριση και το πρωτόκολλο της 5 η Μαΐου του 2010. Οποιαδήποτε ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων θα πρέπει να γίνονται με συμφωνητήρηση αν θέλετε των κανόνων που ισχύουν ε, και στις δύο χώρες διποστασία των προσωπικών δεδομένων η, η κυρία Λίχτεμπέργκερ επέμεινε στην, ε, για την προστασία του περιβάλλοντος. Συμφωνώ μαζί της και όντως θα πρέπει να αναλυφθούν περαιτέρω δράσεις σε σχέση με τη διαχείριση των καυσίμων και τεχνολογία του περιβάλλοντος. Κυρίες και κύριοι, η δουλειά μου ως συγητού ήταν αρκετά δύσκολη. Δεν ήταν δεν εύκολο το πρωτόκολλο αυτό, προσπαθήσαμε να δούμε με ένα ισότομο, ισότιμο τρόπο τα υπέρ και τα κατά του πρωτοκόλλου δεν ε, ξεκινήσαμε πολύ ενθουσιάωδες υπέρ του πρωτοκόλλου αυτού, αλλά μετά από πολλές συζητήσεις καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι καλύτερο θα ήταν να το δεχθούμε το πρωτόκολλο και όχι να το απορρίψουμε. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητώ να υποστηρίξετε και εσείς το πρωτόκολλο αυτό, να υποστηρίξετε το Κοινοβούλιο το πρωτόκολλο αυτό ευχαριστώ ιδιαίτερα τους συνεργάτες μου και τη γραμματεία μου για την πολύτιμη βοήθειά τους. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, τον συνάδελφο Σαζάτα. Είναι σίγουρα σημαντική η συμφωνία αυτή. Θα ήθελα και πολύ θέλω να πάρουν το λόγο. Θα ήθελα να περιορίσω το λόγο των α, σχεδόν εισηγητών. Τρία λεπτά, ο κύριος Ελκαντράου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεσή του. Νομίζω ότι δεν έχουμε και πάρα πολλές ε, εναλλακτικές λύσεις. Ή θα υπερψηφίσουμε ή θα καταψηφίσουμε. Συμφωνία αυτή. Λαμβάνοντας υπόψη την πρώτη συμφωνία που έχει ζηναυτεί εδώ και χρόνια. Το ερώτημα το συγκεκριμένο είναι πώς θα μπορέσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να φτάσουμε στο καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να περιμένουμε, ε, να περιμένουμε κάτι περισσότερο από την Κομισιό. Ε, θα ε, αναλάβει κάποια δέσμευση, θα κάνει στιγμή της κάποια δήλωση η Κομισιό. Θα πρέπει να μας πει ο εισηγητής αν κάτι τέτοιο είναι λογικό. Συμφωνούμε βεβαίως ότι παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα ε, δικαιώματα δεν είναι τα ίδια για τις ε, αεροπορικές μεταφορές για τις ίπα και για μας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να ασκήσουμε κάποια πίεση, χωρίς να θέλω να πω με αυτό ότι θα καταψηφίσουμε την ε, συμφωνία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, προσπαθήσουμε να επιτύχουμε κάτι περισσότερο. Λαμβάνοντας λοιπόν αυτά που είπα υπόψη και αν έχουμε μια κάποια ε, δέσμευση από την Κομισιόν, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. και η ειδική συμβουλευτική επιτροπή που υπάρχει μπορεί να συζητήσει όλα τα θέματα τα σχετικά. για να μπορέσει στο τέλος να προετοιμαστεί καλύτερη δυνατή συμφωνία. Δεν ξέρω αν ε, εμείς ε, εκπροσωπούμεθα σε αυτή την ε, Συμβουλευτική Επιτροπή, αλλά θα έπρεπε να είμαστε ενήμεροι για τις εργασίες του και την πρόοδο που επιτυχάνετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μάιστερ. Ευχαριστώ πρόεδρο. Είναι γεγονός ότι όντως η συμφωνία αυτή είναι δύσκολη. Χτες, όταν ε, γενικά συζητούσαμε για τις συμφωνίες των τομέων των αέριων μεταφορών είχα πει ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και εμείς μετά την, ε, σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την ε, ε, ε υπάρχει πρόβλημα μετάφρασης Πάλι το ίδιο πρόβλημα λέει ο πρόεδρος. Δεν έχουν κάποια μετάφραση. Διερμηνία. Α, εντάξει είναι τώρα. Ωραία, ξαναρχίζω λέει κυρία Μάιστατ. Όταν συζητούσαμε λοιπόν γενικώ ότι για τις εναέρειες μεταφορές είχαμε πει ότι με την θέση ισχύ της ε, ε, συνθήκης της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει περισσότερες αρμοδιότητες και εξουσίες και πρέπει να εξασφαλίσουμε είχα πει εγώ να ίσες ε, ε, ισότιμες αν θέλετε ε, ισότιμα δικαιώματα και στον κόσμο. Ε, ακούμε εδώ τώρα ότι καλύπτουν, καλύπτονται 60% των ευρωπαϊκών ε, αεροπονικών μεταφορών και δεν υπάρχει ε, ισοτιμία και υπάρχουν διακρίσεις. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν λιγότερου πολίτε από ό,τι έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι ότι είναι ο ε, ο μεγάλος εταίρος οι Ηνωμένε Πολιτείες και εμείς οι μικροί ε, και εμείς επανειλημμένα είχαμε παραπονεθεί ότι η Ευρώπη ε, έχει, οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν μικρότερη η πρόσβαση στην αμερικανική αγορά από ότι οι αμερικάνικες στην ευρωπαϊκή. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανεί όλα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να κάπου να ισορροπηθούν καλύτερα τα πράγματα. Όταν άμα μιλάμε για ε, θέση, για συμφωνία, ε, αυτά τα πράγματα είναι προφανή. Αλλά βεβαίως δεν ε, είπαμε ότι Βεβαίω δεν είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολη η συμφωνία αυτή. Το είδαμε και με το SWIFT, το είδαμε και το, με το PNR ότι υπάρχουν κάποια θέματα στα οποία δεν μπορεί να επιβάλλει τη θέση η Ευρώπη. Η Αμερικανοί βλέπουν την προστασία από την τρομοκρατία με πολύ διαφορετικό τρόπο από το βλέπουμε εμείς. Οπότε σίγουρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Σε γενικές γραμμές ε, λέω ναι, α συμφωνήσουμε με τη συμφωνία όπως είπε και ο εισηγητής και ο κύριος αλλά να έχουμε συνέστηση ότι η συμφωνία αυτή είναι έλλειπης θέλουμε παραπάνω πράγματα και έχουμε δικαίωμα να θέλουμε παραπάνω επόμενη φορά λοιπόν θα πρέπει να πάμε να, να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά όχι μοναχά για την πρόσβαση στην αγορά αλλά και για το περιβάλλον και για την ασφάλεια και όλα αυτά. Ευχαριστώ πάντως τον εισηγητή ο οποίος α, είμαι σίγουρη ότι δούλεψε σκληρά για να φτιάξει την έκθεσή του αυτή. Συμφωνώ θα την υπερψηφίσω αλλά ε, κρίμα που δεν πήγαμε παραπέρα. Η κυρία Λίχτενμπέργκερ. Ευχαριστώ πολύ. Άμα συμφωνήσουμε τώρα, το ότι συμφωνούμε μάλλον τώρα με την έκθεση, παρόλο που έχουμε πολλές επιφυλάξεις, θα πρέπει να δούμε ότι η, αυτά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι Αμερικάνοι θα γράψουν τα παλαιότερα των υποδημάτων τους τις επικρίσεις που κάναμε και όλα αυτά που είπαμε στο Πεκίνο. Α, η, η ιστορία αυτή δεν έχει λήξει για μένα η προστασία όχι μόνο του περιβάλλοντος αλλά η προστασία των πολιτών και των καταναλωτών και των επιβατών είναι πάρα πολύ σημαντική και θα έπρεπε να την προασπίσουμε η, αυτά που προτείνουν οι Αμερικανοί και αυτά που θα πρέπει να εφαρμόσουμε εμείς δίχως να έχουμε κάνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε ε, από άλλα θέματα, οικονομικά, πρόσβαση της αγοράς κτλ. Αυτά για μένα είναι ε, δυστυχή πράγματα που συμβαίνουν. Δεν έχουμε εδώ equal footing όπως λέγεται. Δεν διαπραγματευόμαστε στο ίδιο επίπεδο. Δεν θεωρούμεθα ισότιμοι και που θα έπρεπε να θεωρούμεθα. Και καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχουν πολλές πιέσεις. Αλλά για να είμαι ειλικρινής ε, δεν μπορώ να δεν μπορώ να ξεπεράσω τις επιφυλάξεις μου και να υπερψηφίσω. Μιλάμε για σοβαρότατα θέματα που απασχολούν εδώ και χρόνια το Κοινοβούλιο, τα στάνταρ, στάνταρ στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, προστασία των προσωπικών δεδομένων και αυτή η ιστορία με τις νυχτερινές πτήσεις δεν είναι... Ε, ότι σχετίζεται μοναχά με μελλοντικό άνοιγμα της αγοράς. Ήδη, θέλουν να εφαρμοστούν ορισμένα πράγματα. Γι' αυτό είμαι αντίθετη. Και δεν είδα πουθενά στη δική μας την ε, γνωμοδότηση να λέγεται πουθενά, δεν να λέγεται ότι το θέμα των απαγορεύσεων νυχτερινών πτήσεων παραδείγματος χάρη εμπίπτει αποκλειστικά στην εθνική νομοθεσία ε, και σέβεται τις ε, τοπικές συνθήκες. Ε, ε, ε, για να κλείνω δεν μπορώ να συμφωνήσω. Thank you, Chairman. Um, it's been an interesting debate. Well, it's taken... Ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση μας. Πήρε δέκα χρόνια να φτάσουμε στο παρόν στάδιο και περισσότεροι Όσοι είμαστε εδώ, δηλαδή μετά το 99, γνωρίζουν ε, τι ακριβώς συνέβη. Θαύμα λοιπόν. Σωστό λοιπόν λέγεται ότι υπάρχουν ακόμη κάποιες αδυναμίες εδώ, απλώς για τις νυχτερινές ε, πτήσεις. Θέλω να πω ότι είναι θέμα αρμοδιότητας των εθνικών αεροδρομίων εκείνοι αποφασίζουν και δεν νομίζω ότι, έχει κάτι να κάνει εδώ αυτό το θέμα με την συμφωνία με τη Σούζα. Τώρα, έχω κάποια επιφύλαξη με τα ε, θέματα της απασχόλησης. Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι ούτε για το τι συμβαίνει στην απασχόληση τη ΣΥΠΑ, ούτε σε μας. Το να γίνει κάποια αναφορά είναι ένα θέμα, αλλά δεν θέλω να το κάνουμε ολόκληρη ιστορία. Εκεί που νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε τα πράγματα και ξέρουμε ότι έχουμε και εμείς και η Κομισιόν ε, κάτι να πούμε, είναι τι ακριβώς γίνεται με τις ε, επενδύσεις και πού πηγαίνουν τα πράγματα. Πρόκειται για θέματα σημαντικά που πηγαινουν τα πραγματα προκειται για θεματα σημαντικα που εδω και 10 χρόνια. Υπήρξε μια κάποια πρόοδος, το αναγνωρίζω και πιστεύω ότι σωστά μπορούμε να πούμε ότι χρειαζόμαστε μια πιο προσεκτική ε, προσέγγιση, διότι στην Ευρώπη δεν θέλουμε να είναι μονόδρομος ό,τι αποφασίζεται, θέλουμε να υπάρχει αμοιβαία συμφωνία. Τώρα, για το καμποτάζ να φέρουμε. Νομίζω ότι καλά πήγαν τα πράγματα, αλλά το μήνυμα της δικής μας Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να πούμε ότι καλά έγιναν τα πράγματα, κάπως προχωρούν τα πράγματα, προοδεύουν, αλλά χρειάζεται να ε, παίξουμε και εμείς σκληρό παιχνίδι όπως και οι Αμερικανοί για τα θέματα τα οποία προανέφερα και τις αρμοδιότητες μας. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα προοδεύσουμε ακόμη περισσότερο για τα θέματα αυτά προς τα μένα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ. Έγιναν και δύο ερωτήσεις προς την Επιτροπή. Πριν να ολοκληρώσουμε. Θα δώσουμε πρώτα απ' όλα το λόγο στην Επιτροπή για να απαντήσει πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις που έγιναν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ζαζάντα για την έκθεσή του και για το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε. Σωστά είπε αυτά που είπε, διότι λέγει ότι η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να είναι καλύτερη, όντως, θα μπορούσε να είναι καλύτερη, Κυρίως, εάν προέβλεπε ότι για θέματα ελέγχου και ιδιοκτησία θα μπορούσαν τα πράγματα να πάνε πιο γρήγορα και πιο μακριά. Παρουσιάζοντας την εκθεσή του ο κύριος Ζαζάντα επίσης είπε ότι δεν είναι πάντα δυνατόν να επιτύχουμε αυτό το οποίο επιθυμούμε. <laughs> Λαμβάνοντα και υπόψη το γεγονό ότι ο εταίρο μα θα πρέπει αυτό το οποίο επιζητούμε εμεί επίση να το αποδεχθεί. Όντω υπάρχει μια κατάσταση ανισορροπία σε θέματα ιδιοκτησία και ελέγχου. Αν συγκρίνουμε τους κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ΣΥΠΑ. Δεν είναι τυχαίο και γι' αυτό το λόγο εξάλλου οι, οι υπηρεσίες αερομεταφορών τα καλύπτονται από τον ΚΑΤΣ. Ξέρω ότι έχουν τρομερέ δυσκολίε οι Αμερικανοί. Η... Πενθύμησε την κατάσταση ο εισηγητή που έχει ως εξή. Ή θα αποδεχθούμε μία συμφωνία που τελικά προβλέπει ότι κάποια μέρα θα φτάσουμε μέχρι τέλους σε θέματα ελέγχου τη ή δεν θα έχουμε καμία συμφωνία. Το να μην υπάρξει καμία συμφωνία, τι σημαίνει για μας. Ότι δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί πρόοδο σε κανένα από τα σημεία που θεωρούμε σημαντικά και όπως είπε και ο κύριος Ζαπάντα, προστασία των καταναλωτών, περιβάλλον, ασφάλεια βεβαίως και κοινωνική πτυχή του όλου θέματος. Και βεβαίως έχουμε και την Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή που με την εργασία που επιτελεί θα επιτρέψει κάποια μέρα στον τομέα αυτό να απελευθερωθεί πλήρως. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Παρ' όλα αυτά, η συμφωνία αυτή πιστεύω ότι αποτελεί μια βάση σταθερή από την οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε για να ευρεώσουμε ακόμη περισσότερο τις ε, υπερατλαντικές σχέσεις μας για τις στον τομέα των αερομεταφορών. Και βεβαίως εμείς από την Κομισιό υπολογίζουμε σε εσά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το Αμερικανικό Κογκρέσο επίσης να σκεφτεί <coughs> το θέμα αυτό. Της ιδιοκτησίας και του ελέγχου. Εξάλλου, αυτό είναι και το αντικείμενο των επισκέψεων που γίνονται στακτά διαστήματα από μέλη της Επιτροπής σας και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες επισκέψεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε την πρόθεση να οργανώσουμε με τη ΣΥΠΑ ένα φόρουμ για τις επενδύσεις όπως οργανώσαμε και για θέματα ε, απασχόλησης πέρσι, που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε για κάποια θέματα και θέματα τα οποία είναι κεντρικά και σημαντικά η συμφωνία αυτή. Και βεβαίως θα κληθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει στο φόρουμ αυτό που θα οργανώσουμε. Κύριε Ελκαντράουι. Αναφέρατε μία τρίτη φάση, μία τρίτη φάση διαπραγμάτευσης μάλλον. Είναι δυνατόν, είναι επιθυμητό να γίνει κάτι τέτοιο. Εμείς με τους Αμερικανούς νομίζω ότι φτάσαμε μέχρι σε σχάτων όσον αφορά σήμερα τι μπορούμε να επιτύχουμε. Επαναλαμβάνω, η συμφωνία προβλέπει σε διαδοχικές φάσεις ότι κάποια μέρα θα επιτύχουμε την πλήρη απελευθέρωση του τομέα αυτού. Δεν είμαι σίγουρος ότι μια νέα συμφωνία θα έχει να προσθέσει κάτι συμπληρωματικό, δεδομένου ότι σήμερα έχουμε τα μέσα να φτάσουμε, όπως σας λέω, μέχρι σε Βεβαίως χρειάζεται ακόμη να γίνει πολλή δουλειά για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συμφωνία σε θέματα ιδιοκτησίας κυρίως και ε, ελέγχουμε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και βεβαίως είναι απολύτως νόμιμο να εκφράζονται κάποιες ε, ανησυχίες ας πούμε παράπλευες, σε σχέση με την πλήρη απελευθέρωση των αερομεταφορών που είναι το κεντρικό θέμα αυτής της συμφωνίας. να υπάρχουν αυτές οι ανησυχίες που αφορούν βεβαίως την προστασία των προσωπικομένων την προστασία του περιβάλλοντος. Χθε, στα πλαίσια της συζήτηση που έγινε εδώ για την έκθεση του κυρίου Σίμψον, είπα ότι οι συμφωνίες στον τομέα της αεροναυπλίας δεν μπορούν αυτές να ρυθμίσουν κάποια εγκάρσια θέματα. Αντιθέτως όμως, μπορούν να συνεισφέρουν στο να χειριστούμε όλα αυτά τα θέματα με τον καλύτερο δυνατικό τρόπο, όπως φερειπίν η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σίγουρα μπορεί κανείς στα πλαίσια μιας γενικής συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Σίγουρα, σίγουρα. Με το περιβάλλον. Το θέμα του θορύβου που ανέφερε η κυρία Λίχτενμπέργκερ της συγχωρήπανση. Δεν θα γίνει τίποτε, εάν μπορώ να το πω αυτό, δεν θα γίνει τίποτε όσον δεν αλλάξουμε στα πλαίσια της συναπόφασης, το Συμβούλιο και εσείς δηλαδή, την οδηγία για την ηχορύπανση. Και όπως σας είπα και επαναλαμβάνω, εσείς έχετε την τελευταία λέξη για αυτό το θέμα. Τώρα, στα πλαίσια της ε, θέσης ίσχυ αυτής της συμφορίας, μπορούμε να συζητήσουμε με τους Αμερικανούς το προβλέπουν για τα δικαιώματα των επιβατών. Διότι υπάρχει για τα δικαιώματα των επιβατών σχετική αμερικανική νομοθεσία που θα μπορούσε να έρθει σε αντιπαράθεση με τη δική μας νομοθεσία. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της συμφωνίας θα μπορούσαμε να επιστήσουμε την προσοχή των ήπα σε δυσκολίες που θα μπορούσαν να ανακύψουν ενδεχομένως. Αυτά ήθελα να απαντήσω κύριε Πρόεδρε, για να απαντήσω στις ανησυχίες και στα σχόλια που έκαναν κάποιοι συναδελφοί σας και βεβαίως θα σας ενημερώνουμε για την πρόοδο όσον αφορά αυτή τη συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε τι είχε να πει η Κομισιόν. Επίσης, ε, θα ήθελα να μας πείτε κάτι για μια δήλωση που είπαμε θα θέλατε να κάνετε ως Επιτροπή στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Το θέμα που τέθηκε αφορά μια δήλωση για την τρίτη φάση διαπραγμάτευσης. Απάντησα ότι Ίσως αυτός δεν θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε στη σχέση μας με τις είπαμε. Με αυτή τη συμφωνία <coughs> έχω την εντύπωση ότι πήγαμε όσο πιο μακριά μπορούσαμε στα θέματα που συζητούμε με τους Αμερικανούς εταίρους μας. Αντιθέτως, είναι σημαντικό, θα έλεγα, και με την ε, συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προχωρήσουμε για τη συγκεκριμένη εφαρμογή αυτής της εφαρμογής. Διότι ελπίζουμε ότι κάποια μέρα θα υπάρχει μεγάλο ποσοστό ιδιοκτήτων αεροπορικών ε, ιδιοκτητριών αεροπορικών εταιριών των, ε, της Ευρώπης στη ΣΥΠΑ ελπίζουμε βεβαίως και το αντίθετο μπορεί να συμβεί. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν χρήσιμο να ζητήσουμε ε, να μας ανατεθεί από το Συμβούλιο εντολή διαπραγμάτευσης νέας συμφωνίας για θέματα ιδιοκτησίας και ελέγχου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση τώρα. Πριν να δώσω το λόγο στον εισηγητή. Κύριε Λίχτενμπέργκερ να μην ξανανοίξουμε συζήτηση. Δεν θα αναφερθώ επί της ουσίας, παρόλο που ο πειρασμός είναι μεγάλος. Αυτά που είπε η Κομισιόν δεν ήταν ε, καθησυχαστικά. Αλλά η Κομισιόν λέει ότι δεν θέλει να κάνει δήλωση. Εμείς λέμε παρόλο που δεν θεωρούμε καλή την πρόταση, παρόλα αυτά θα την υπερψηφίσουμε. Ρωτώ, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα ψήφισμα ή ένα κάποιο ε, κείμενο το οποίο να περιλαμβάνει αν θέλετε τις επικρίσεις ε, που ακούστηκαν για τη συμφωνία αυτή διότι αλλιώς θα μας κροϊδεύουν οι Αμερικάνοι maken eh, Μήπως θα μπορούσατε να καταλήξετε στα τελευταία σας τελικά σας συμπεράσματα και να μας δώσετε μια κάποια ένδειξη για το τι πρόκειται να γίνει. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρα. Έχουμε εξάγει τα συμπεράσματα τα οποία βρίσκονται ήδη στο έγγραφο. Υπάρχει μια έκκληση για περαιτέρω βήματα τα οποία θα πρέπει να κάνουμε. Η Κομισιόν θα πρέπει να διαπραγματευτεί τα επόμενα στάδια της συμφωνίας και υπάρχουν και άλλα κεφάλαια στα οποία θα πρέπει να υπάρξει μια κάποια πρόοδος, ελευθεροποίηση των ανοίγμα των πτήσεων, καλύτερο συντονισμός ε, ε, των στρατηγικών όσον φορά επίσης ε, τα δικαιώματα των επιβατών, δηλαδή μεγαλύτερη προστασία των επιβατών ουσιαστικά. Και όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο. Και επίσης απευθύνουμε μια έκκληση στην Κομισιό να προχωρήσει παραπάνω μας δυσαρεστεί λίγο το γεγονός ότι η Κομισιό είναι τόσο ευχαριστημένη από το έργο της, διότι ναι, μεν είναι καλά όσα έχουν γίνει, όμως θα πρέπει να είμαστε κάπως πιο φιλόδοξη Δεν έχουμε υλοποιήσει όλα μας τα όνειρα εδώ. Έχουν γίνει απλώς κάποια βήματα. Βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση μεν και ίσως ε, να υπάρχει κάποια μέρα να δημιουργηθεί ο, ο, ο, ο ενιαίος παγκόσμιος ουρανός. Ξέρω ότι αυτό που μας ε, απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι ο ευρωπαϊκός ουρανός, αλλά ε, νομίζω ότι το όραμά μας πρέπει να είναι να έχουμε τους, ε, τον ενωμένο παγκόσμιο εθέρα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ μιλάμε για το 60% της παγκόσμιας, ε, των παγκόσμιων αεροπορικών ε, μεταφορών. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και θα πρέπει να υλοποιήσουμε τα όνειρά μας κάποια στιγμή. Υπάρχει αυτή η μεικτή επιτροπή η οποία θα αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα και υπάρχουν κάποιες προβλέψεις ε, όσον αφορά τι είναι συνεργασία, η οποία γίνεται εφικτή ούτως ή άλλως. Αλλά θα, ήθελα η αλλως αλλα θα ηθελα η κομισιο να, να συνειδητοποιήσει ότι εμείς αμέλη του Κοινοβουλίου θέλουμε όλα αυτά να γίνουν νωρίτερα, όχι αργότερα. Τώρα, κοιτάξτε, μην αρχίσουμε πάλι να δίνουμε το λόγο σε όλους ε, όσους, πήραν, όσους μίλησαν. Το πρόβλημα είναι τι θα γίνει με την συμφωνία αυτή. Θα την καταπιούμε όσα έχει. Βέβαια υπάρχει ε, και δυνατότητα για το ψήφισμα ε, με ε, η υποβολή τροπολογιών μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου. 20 Φεβρουαρίου θα συζητηθεί στην... Ε, ε, Φεβρουαρίου θα συζητηθεί στην Επιτροπή μας και μετά θα περάσει από, το, Βέβαια θα πρέπει να δούμε στο ψήφισμα τι θα συμπεριλάβουμε. Μήπως εκεί μπορούμε να ασκήσουμε μια μεγαλύτερη πίεση. Δηλαδή θα πρέπει και ο εισηγητής να συνεργαστεί με τους ε, συναδέλφους έτσι ώστε να ε, γίνει πιο δυνατό αν θέλετε το, το ψήφισμα. Λοιπόν, σας ζητώ να συζητήσετε ε, περισσότερο με τους συναδέλφους να είναι πιο ισχυρό το ψήφισμα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα. Τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα μας που αφορά τη Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών με την βόρεια γείτονα, με την γείτονα προς βορρά του ΗΠΑ, με τον Καναδά, η συγγήτρια, κυρία Τικάου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η, η έκθεση την οποία συζητάμε τώρα αφορά την ε, Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά. Είναι μια συμφωνία πλαίσιο και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή συμφωνία, διότι οι διατάξεις της ε, είναι ισορροπημένες, ε, δηλαδή και τα δύο μέρη έχουν τα ίδια δικαιώματα και ήθελα να πω ότι πριν ε, δημιουργηθεί αυτή εδώ η συμφωνία είχαμε 19 διμερείς συμφωνίες ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, αποφάσισε ότι κάποιες από αυτές τις ε, διατάξεις των διμερών συνθήκων δεν ήταν ε, ε, συμβατές με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, εξού και εδόθη ε, η ε, να είδωσε εντολή στην, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευτεί, να προτείνει και να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με την ε, ενιαία συμφωνία με τον Καναδά. Η, θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή συμφωνία. οι, ε, οι επενδύσεις θα ρέουν χωρίς καμία, κανέναν εμπόδιο και ε, μπορούν οι αεροπορικές εταιρείες να λειτουργούν και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού κανονικά, ακόμα και στο εσωτερικό και στην εγχώρια αγορά. Η συμφωνία αυτή αναγνωρίζει ε, βέβαια ότι δεν μπορούμε να έχουμε απόλυτα ο άνοιγμα ε, των, για τις επενδύσεις από την αρχή και θα υπάρχουν τέσσερα στάδια στη συμφωνία. Το πρώτο στάδιο ξεκινά όπου το, ε, ε, εκεί που το ποσοστό της ξένης ιδιοκτησίας περιορίζεται στο 25%, το δεύτερο στάδιο στο 49% των μετοχών, το τρίτο στάδιο ξεκινά μόλις τα δύο μέρη επιτρέψουν στους επενδυτές να ιδρύουν και να ελέγχουν νέες αεροπορικές εταιρείες στην αγορά του άλλου μέρους και το τέταρτο στάδιο που είναι και το τελευταίο και εκεί παραχωρούνται πλήρη δικαιώματα εκτέλεση δρομολογιών και μέσα και πέραν των αντίστοιχων αγορών. Επίσης υπάρχει μια σταδιακή, αν θέλετε, κλιμάκωση των δικαιωμάτων αυτών. Επίσης στείλονται θέματα όπως η ασφάλεια, τα δικαιώματα των ε, επιβατών, ε, ανταγωνισμός και οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν έτσι ώστε να εξασφαλίσουν και ένα χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο θα υπάρξουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών και την, τα δικαιώματα αποζημίωσης. Επομένως βλέπετε ότι υπάρχουν μέτρα ε, που ενισχύουν τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση που δεν τους επιτραπεί να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο. Και αυτή η συμφωνία είναι πιο φιλόδοξη από αυτήν ε, ε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές. Ε, βέβαια στην κοινωνική ε, διάσταση δεν είναι τόσο φιλόδοξη. Γι' αυτό είναι σημαντικό η Κομισιό να χρησιμοποιήσει αυτή την συμφωνία και κυρίως τον, τις αρμοδιότητες που έχει για να ζητήσει από την Μικτή Επιτροπή να υπάρξει σε διεθνές επίπεδο μια περαιτέρω προώθηση όλων αυτών των κοινωνικών δικαιωμάτων. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Ήταν ε, σαφής και σύντομη η παρουσίασή σας και απευθύνομαι στην, ε, στους συναδέλφους του κ. Κούς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για το σχέδιο σύστασης. Πράγματι πράγματι εδώ λέγονται όλα αυτά που χρειάζεται να πει κανείς για, αυτό το για αυτή τη συμφωνία εγώ θα έλεγα κιόλα το σχέδιο αυτό συμφωνία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ω υπόδειγμα, αν θέλετε, και για άλλε συμφωνίε όπω παραδείγματο χάρη είναι αυτή ε, με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Αναφέρεται και μια τέταρτη φάση. Ε, εδώ, αν κατάλαβα καλά, δεν ε, ε υπάρχει καν ο φόβο να αναφερθεί στην τελευταία και τέταρτη φάση, το καμποτάζ δηλαδή ένα πλήρε άνοιγμα των αγορών την κοινωνική πτυχή θα μπορούσαν να γίνουν ορισμένε παρατηρήσεις ε, συμφωνώ με αυτές που έγιναν συμφωνώ επίσης με τα σχόλια που έγιναν για την ασφάλεια ε, Συμφωνώ με αυτό που λέγεται στο κείμενο ότι θα πρέπει ίσως να αναθεωρηθούν κάποια πρότυπα ασφάλειας ε, που ισχύουν αυτή τη στιγμή για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα της αναγνώρισης και της απλούστευσης των, ο, της, εκμε, της χρήσης αν θέλετε ε, της εφαρμογής και από την πλευράς χρηστών ε, θα ήταν πραγματικά ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα το να αναγνωρίσει κανείς αμοιβαίως τα πρότυπα, τα πρότυπα που ισχύουν συμφωνώ λοιπόν ε, σε γενικέ γραμμές με την ε, έκθεση, με τη σύσταση, ε, υπερψηφίζω. Ναι. Ε, κυρία Μάισνερ για τους φιλελεύθερους ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε ευχαριστώ και την κυρία Τίκαου για την έκθεση. Δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα μετά από αυτά που ελέγχθησαν. Όλα τα σημαντικά έχουν μπει στην έκθεση. Συμφωνώ, συμφωνώ με την έκθεση αυτή. Το σου το μάλλον που συμφώνησα προηγούμενα είπαμε ε, ότι θα υπερψηφίσουμε και τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να, εδώ υπάρχουν πολλά πολλά καλύτερα πράγματα από αυτά που υπάρχουν συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ καλή συμφωνία λοιπόν με τον Καναδά. Υπέρ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λίχτεμπεργκερ. Ναι, θα μπορούσα να συμφωνήσω κι εγώ στο γεγονός ότι τούτη η συμφωνία είναι πράγματι πολύ πιο εξισορροπημένη από την προηγούμενη που συζητούσαμε. Εμείς ως Ευρωπαίοι και Ευρωπαίες θα πρέπει να πούμε πολύ πιο ξεκάθαρα ότι συναντιόμαστε ή συζητούμε σε ισότιμο ίσο επίπεδο. Δεν είμαστε αφεντικό και υπηρέτης ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να φανταστεί κανείς πάνω σε αυτές τις γραμμές. Είμαστε ισότιμοι στις συμφωνίες αυτές και αυτό πρέπει να φαίνεται παντού και στην κοινωνική πτυχή, στις κοινωνικές διατάξεις ε, που δεν φαίνεται και τόσο πολύ βέβαια αλλά τέλος πάντων σε γενικές γραμμές η συμφωνία αυτή είναι καλή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για να γίνουν τα περαιτέρω βήματα που είναι αναγκαία να γίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπρέκπολ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να μιλήσω και σαν, αυτό θέλω να πω, σαν πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Καναδά. Όπως ε, και οι περισσότεροι συναδέλφοι εδώ, έχουμε κάποια προβλήματα με αυτή τη συμφωνία. Θα ήθελα όμως να κάνω και κάποιες παρατηρήσεις, ε, διότι και σε αυτήν, ε, αυτή η συζήτηση αλλά και άλλες συζητήσεις ε, ε έδειξαν κάποια προβλήματα και απευθύνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ένα πράγμα σε, γενικό, σε ένα γενικότερο πλαίσιο ε, ισχύει, η Κομισιόν θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κάτι δεδομένο. Δηλαδή ότι είμαστε εδώ απλώς και μόνο για να επικαιρώνουμε τις συμφωνίες που ε, κάνει εκείνη. Όμως ε, το Κοινοβούλιο έχει να παίξει ένα πολύ πιο ουσιαστικό ρόλο στον καθορισμό αυτών των συμφωνιών και η Κομισιόν θα πρέπει να το συνειδητοποιήσει αυτό και θα πρέπει να ενημερώνει ε, από την αρχή μέχρι το τέλος ε, το κοινοβούλιο αυτό για τις συμφωνίες ε, που διαπραγματεύεται και όχι μονάχα στον σεναρίες μεταφορές σε, έναν μεγάλο σε ένα μεγάλο αριθμό τομέων. Για το SWIFT παραδείγματο χάρη η Κομισιό θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα κάποιο βάρος και θα πρέπει να το διαβουλεύει, θα πρέπει να το, να, να το ενημερώνει τουλάχιστον. Τέλος πάντων, θα ήθελα να καλωσορίσω βέβαια την συμφωνία αυτή, την οποία θεωρώ θετική και πιστεύω ότι... Ε, παρακολουθήσαμε ε, την ε, συμφωνία αυτή και εντάσσεται η συμφωνία αυτή στο γενικότερο πλαίσιο των ε, συμφωνιών με τον ε, Καναδά. Βέβαια, γιατί αυτή η συμφωνία δεν διαπραγματεύτηκε εν κενό, ε, εντάχθηκε στο γενικότερο πλαίσιο των εμπορικών σχέσεων και συμφωνιών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στον, στον Καναδά. Οι δύο θέματα τα οποία τα έθιξαν ακροθυγώς οι συνάδελφοι. Το ένα είναι η ασφάλεια των αεροδρομίων. Όλοι θέλουμε να πετύχουμε ε, αυτό. Όμως δεν μπορούμε να ε, εξετάσουμε εδώ τον Καναδά ε, απομονωμένα, διότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της κίνησης από την ευρωπαϊκή κοινότητα στην, στον Καναδά περνάει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως θα πρέπει να λύσουμε το θέμα του transit, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούμε να το λύσουμε το πρόβλημα είναι ένα τρίγωνο, δηλαδή εάν περάσεις από τον Τορόντο ή από, τον, από το Μόντρεαλ και τα μπορείς να έχεις ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας. Αν αυτό όμως γίνει, το τράνζιτ είναι από, τον, από τη Ουάσιγκτον ή από τη Νέα Υόρκη ή οπουδήποτε άλλο, είναι άλλο, το, άλλη κατάσταση και ναι, μεν καλωσορίζω τα βήματα προόδου αυτής της συμφωνίας, όχι μονάχα στα θέματα ασφάλειας, αλλά και σε γενικότερους όρους ανοίγματος της αγοράς, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν μπορούμε τον Καναδά να τον εξετάσουμε απομονωμένα από, τις υπόλοιπες, από την υπόλοιπα Βόρεια Αμερική. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ακούστηκαν πολλές ερωτήσει ε, στην Κομισιόν και οι οποία θα πρέπει να απαντήσει. Κοιτάξτε, ευχαριστώ την εισηγήτρια για την έκθεση και για την ε, θετική εκτίμηση που έκανε, θετική αξιολόγηση που έκανε ε, για αυτή τη συμφωνία, κάτι το οποίο νομίζω ότι συμμερίζεται όλη η Επιτροπή. Και αυτό ευθυγραμμίζεται με το γεγονός ότι η συμφωνία αυτή είναι μάλλον και σίγουρα θα έλεγα η καλύτερη που έχουμε μέχρι τώρα. Και ο κύριος Γκρόσο πολύ σωστά είπε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μοντέλο. Ε, θα θέλαμε όλες μας οι συμφωνίες να ακολουθήσουν το, τα πρότυπα της συμφωνίας ε, με τον Καναδά. Αυτό όμως δεν είναι πάντα εφικτό. Το είδαμε και στην περίπτωση της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία ήδη έχει επιφέρει καρπούς, διότι ο η καναδική νομοθεσία που επιτρέπει να περάσουμε από το 25% στο 49% των μετοχών ε, που ανήκουν σε ξένους ε, ε, επενδυτές έχει γίνει, των μετοχών των καναδικών εταιριών δηλαδή, έχει ήδη περάσει. Θα πρέπει να δημοσιευθεί βέβαια η νομοθεσία, ο νόμος αυτός. Επομένως ήδη είμαστε στην, ε, στο δεύτερο στάδιο. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αποκτήσουμε νέα δικαιώματα ε, κυκλοφορίας. Επομένως έχει ξεκινήσει η διαδικασία μέσα στα πλαίσια αυτής της ε, συμφωνίας. Και αυτό είναι κάτι που μας χαροποιεί. Είναι αληθές βέβαια ότι σε ένα θέμα, ένα θέμα, σε ένα θέμα δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε όσο θα θέλαμε και είναι το θέμα της απασχόλησης, το άρθρο 19 αυτής της συμφωνίας, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι η διαπραγμάτευση του, για αυτό το άρθρο ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ε, συναντήσαμε μεγάλη αντίσταση από πλευρά των Καναδών για να συμπεριλάβουμε μία διάταξη για την απασχόληση την δεχτήκανε τελικά, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ε, κάθε φορά που είναι απαραίτητο θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την διάταξη της συμφωνίας για όλα τα υπόλοιπα στοιχεία και δεν θα τα αναφέρω τώρα. Η κυρία Τικάου έκανε μια παρουσίαση ε, πλήρη. Ε, είχαμε μεγάλη πρόοδο. Ένα σημείο, ένα θέμα το οποίο έθιξε ο κ. Μπαγκμόν είναι η ασφάλεια βέβαια. Ήδη έχουν γίνει, έχει γίνει μια πρόοδος και απτή πρόοδος το έλεγα ε, και ε, θέλουμε να, να εφαρμόσουμε αυτό το οποίο ονομάζεται One Stop Security. Βέβαια σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα προβλήματα που δημιουργεί το transit μέσω των ΗΠΑ. Όμως ε, ήδη στο, με τον Καναδά, στο σημείο αυτό έχουμε πετύχει πρόοδο. Αυτά ήθελα να υπογραμμίσω πρόεδρε από πλευράς της Κομισιόν και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά την κυρία Τικάου για την έκθεσή της. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος, για τις απαντήσεις σας. Η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους. Νομίζω ότι πρόκειται για μια παραδειγματική, υποδειγματική ε, συμφωνία που θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για επόμενη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ελπίζω να την υποστηρίξετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. όπως και για τις επόμενες συμφωνίες, ε, μπορούμε να τις υιοθετήσουμε, να τις απορρίψουμε. Επίσης, μπορούμε να υιοθετήσουμε μια, ένα ψήφισμα 2 Φεβρουαρίου προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, 28 Φεβρουαρίου η συζήτηση στην ε, Επιτροπή μας και θα περάσει από την Ολομέλεια του Μαρτίου. Ευχαριστώ κύριε Τικάου και τους άλλους ομιλητές βέβαια. Περνάμε στο επόμενο σημείο, Συμφωνία Ευρωπαϊκής Κοινότητας Βραζιλίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Η κυρία Τικάου πάλι. Η συμφωνία με την Βραζιλία αφορά την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Είναι διαφορετική η συμφωνία αυτή από την συμφωνία πλαίσιο την οποία μόλις συζητήσαμε. Η συμφωνία αυτή με την Βραζιλία υπογράφηκε στις 14 ε, Ιουλίου του 2010 και δεν έχει τεθεί σε προσωρινή εφαρμογή. Αυτό χρειάζεται απόφαση του Συμβουλίου. Μέχρι ολοκληρωθεί η συμφωνία, η Βραζιλία έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες πιστοποίησης προϊόντων με έξι μόνο κράτη-μέλη. Αυτές οι διμερείς συμφωνίες θα τερματιστούν την ημέρα που θα τεθεί σε ισχύ ή εν συμφωνία. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι καλό, διότι παγιώνει την αμοιβαία αποδοχή των πορισμάτων πιστοποίησης σε όλα τα πεδία της αξιοπλοείας για όλα τα κράτη-μέλη. Ε, επίσης, δίνεται δυνατότητα τροποποίησης των παραρτημάτων ε, της συμφωνίας αργότερα. Και θα θέλαμε να ζητήσουμε από την Κομισιό να κρατάει το Κοινοβούλιο ενήμερο, ενήμερο όταν πρόκειται να αλλάξει τα σημαντικά από αυτά τα παραρτήματα. Ε, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να προλάβουμε την ε, ε, επικάλυψη σε αξιολογήσεις, δοκιμές και ελέγχους σε σημαντικά, σε επισημαντικών κανονιστικών διαφορών και να χρησιμοποιείται το σύστημα πιστοποίησης και από τα δύο μέρη για να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άλλου μέρους. Η συμφωνία ακολουθεί σε γενικέ γραμμέ τη διάρθρωση των ε, υφισταμένων διμερών συμφωνιών για την ασφάλεια των ε, αερομεταφορών Ε, η συμφωνία αυτή διατυπώνει υποχρεώσει και παρέχει μεθόδου συνεργασία ώστε η αρχή εισαγωγή να μπορεί να εκδίδει τα δικά τη πιστοποιητικά για αεροναυτικά προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμό, χωρίς να χρειάζεται να επαναλάβει όλες τις αξιολογίες που έχει πραγματοποιήσει η αρχή εξαγωγής και ολοκληρώνω λέγοντας ότι υπάρχει ευελιξία, υπάρχει η απαραίτητη ευελιξία να αντιδράσουμε άμεσα σε τις περίπτωση που εχει πραγματοποιησει η αρχη εξαγωγη και ολοκληρωνω λεγοντα προβλήματα ασφάλειας. και πιστεύω ότι η συμφωνία αυτή θα ωφελήσει σημαντικά και τις βραζιλιάνικες εταιρείες αλλά και τις ευρωπαϊκές διότι ε, εισάγει συντομότερες και απλούστερες ε, και πιο οικονομικές διαδικασίες έγκρισης προϊόντων και αμοιβαία αποδοχής των πορισμάτων πιστοποίησης. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα να ακούσω τους συναδέλφους στα... για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Τικάου. Σας ευχαριστώ για την ε, παρουσίασή σας ε, που ήταν ε, ιδιαίτερα ποιοτική. Απευθύνομαι τώρα στις εκπροσώπους των ομάδων. Τρία λεπτά αναομιλητή. Ευχαριστώ, πρόεδρα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι η συμφωνία μεταξύ Βραζιλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα σημαντικό θέμα σε θέματα ασφαλείας των αεροναυτιλίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για μας και με συμφωνίες προστίτητες χώρες και για την ασφάλεια στον ευρωπαϊκό χώρο. Η... Ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπήρχαν προβλήματα, τώρα δίδονται νέες δυνατότητες και γίνονται νέες επενδύσεις για να ανοίξουν. Παρακαλώ, λέει ο πρόεδρος. Υπάρχει πάλι κάποιο πρόβλημα τη διερμηνία. Oh. Het punt, het punt schijnt te zijn dat er geen Portugees is. Ik Ik weet even niet wat dat technisch betekent, maar ik... Αυτό δεν δουλεύει κανεί. Α, κατάλαβα. Ενώ εγώ άρεσα. Εσύ ναι. <laughs> Ε, beste mensen, we hebben een probleem. Eh. Έχουμε ένα πρόβλημα, λέει ο πρόεδρο. Διότι δεν προβλέπονται τα πορτογαλικά στην ε, συνεδρίαση αυτή. Άρα δεν μπορείτε να μιλήσετε αυτή τη γλώσσα. Τα Ολλανδικά σας όμως είναι πολύ καλά. Αν θέλετε συνεχίστε στα Ολλανδικά. Μια στιγμή, μια στιγμή. Οι διερμηνεί λένε ότι δεν έχουμε Πορτογαλικά.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 αλλά θα μιλήσω αγγλικά, αλλά θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ. Θέλω κι εγώ να μιλώ τη μητρική μου γλώσσα, δεν είμαι ο μόνος Πορτογάλος, υπάρχει και ένας αναπληρωτής, θα ήθελα να παρακαλέσω δηλαδή την Κομισιό, ενώ θέλει να πει το Κοινοβούλιο, ο κύριος Τεσέρα να το λάβει υπόψη ε, την δεν ξέρω τι συνέβη, λέει ο Πρόεδρος. Λαμβάνουμε υπόψη την δήλωσή σα. Συμφωνώ με αυτά που είπατε. Θα δούμε σε επίπεδο, όχι κομισιόν, συγγνώμη, σε επίπεδο τη δική μα επιτροπή τι μπορεί να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε. Θα δούμε τι θα μπορούμε να κάνουμε. Τέλο πάντων, θα κάνω μια προσπάθεια ενδεχομένω να μιλήσω Ολλανδικά. Λοιπόν, θα τα πω αγγλικά. Επειδή ο χρόνο είναι πολύτιμο και να μην μακρηγορούμε, θα ήθελα να πω το εξή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Τσικάου, για την εξαιρετική εργασία της. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι η συμφωνία αυτή είναι εποφελής και για τα δύο μέρη, και για τη Βραζιλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορώ να πω στην Επιτροπή σας ότι χθε δείπνησα με τον πρέσβη της Βραζιλίας και τόνισε δύο πράγματα πολύ σημαντικά για τη Βραζιλία. Πρώτα απ' όλα, συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ και δεύτερον, οι δύο συμφωνίες για τις ε, αερομεταφορές που εκκρεμούν ακόμη στο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο. Επίσης και για μας είναι υποφελή συμφωνία, διότι η Βραζιλία θα γίνει κάποια στιγμή η πιο σημαντική η οικονομία αναπτυσσόμενη στον κόσμο και είναι ο δέκατος εταίρος εμπορικός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία αυτή έχει πολύ άριθμα σημεία τα οποία είναι εποφελή για όλους και βεβαίως είναι σημαντικότητα για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Διότι εδώ αναγνωρίζεται η πιστοποίηση, ενισχύεται η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ Βραζιλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικατοπτρίζει το πνεύμα που επικρατεί στον τομέα της πολιτικής απορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από διαδικαστικής πλευράς. Θα πω ότι λυπούμε που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει σε πολύ ε, πολύ αργά αν θέλετε στην όλη διαδικασία. Και, τονίζω και πάλι την πρόκειται για μια συμφωνία πολύ σημαντική και για τους δύο εταίρους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ε, ευχαριστώ και για τις ε, γνώσεις σας, τις γλωσσικές, λέει ο Πρόεδρος. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη για να κερδίσουμε το χρόνο που χάσαμε σήμερα με όλες τις τεχνικές, όλα τα τεχνικά προβλήματα. Θα πω απλώς ότι συμφωνώ με την... θα ψηφίσω υπέρ της συμφωνίας αυτής αν θέλετε, αλλά θα μπορούσαμε και εδώ να έχουμε κάποια ακόμη καλύτερα πράγματα από αυτά που αναφέρονται. Αλλά είμαι υπέρ. Τέλεια λέει ο πρόεδρος. Πάρα πολύ ωραία. Άμα όλοι μιλούν έτσι, τότε θα προλάβουμε να πάμε και για καφέ. Λίχτενμπεργκεν, θέλω να ρωτήσω κάτι, τι, δυστυχώς. Ε, στη Βραζιλία είχαμε προβλήματα ασφάλειας ε, με τις απαιτήσει, όχι ασφάλειας με την έννοια του security, ασφάλεια με την έννοια του safety. Και είχαμε πει ότι θα μελετηθούν αυτά και θα επιληθούν πριν να κάνουμε ένα επιπλέον βήμα. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν την Επιτροπή τι έγινε σχετικά. Ναι βεβαίως λέει ο ο πρόεδρος θα ρωτήσουμε την Κομισιόν Τζάκι Φώστερ Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή κυρία Πρόεδρε. Έκανε την, την εισηγήτρια, έκανε εξαιρετική δουλειά. Επελήθησαν τον εισηγητή. πολλά προβλήματα που είχαμε με τη Βραζιλία στο παρελθόν ε, και νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και στην Κομισιόν και στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Η Κομισιόν τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να απαντήσει την ερώτηση τη κυρίας Λίχτενμπέργκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Τικάο για την ε, έκθεσή της ε, και το, για το συμπέρασμα ε, στο οποίο κατέληξε. Χαιρόμαστε γιατί και η, η Κομισιόν χαίρεται, διότι κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα, όπως και με την συμφωνία με τον Καναδά όσον αφορά την ασφάλεια. Κατανοώ επίσης ε, και τις ερωτήσεις ε, τις ερωτήσεις για τη συμφωνία αυτή. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια γενικότερη συνένεση Όπως και με τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και εδώ θέλουμε να υπάρχει η αμοιβαία αποδοχή των πιστοποιητικών και όσον αφορά την ναυσιπλοεία, την αρχική ναυσιπλοεία, δηλαδή την πιστοποίηση των προϊόντων, των αεροναυτικών προϊόντων και ε, των ε, οργανισμών σύλληψης και παραγωγής αυτών των προϊόντων, αλλά θέλουμε και την αμοιβαία αποδοχή των πιστοποιητικών της συνεχούς ναυσιπλοείας ε, που συνδέονται με την λειτουργία των αεροσκαφών αλλά και τη συντήρηση των αεροσκαφών, όπως επίσης και την συντήρηση των ε, ανταλλακτικών τους. Όλα αυτά είναι ένα πράγμα. Αλλά πιστεύουμε ότι με τη συμφωνία αυτή ανοίγουμε το δρόμο ε, σε μια στενή συνεργασία με την Βραζιλία, που δεν χρειάζεται να στο το υπενθυμίσω, είναι η τέταρτη παραγωγός σε αεροναυτικά προϊόντα στον κόσμο. Και θέλουμε η συνεργασία αυτή να διευρυνθεί πέραν της αμοιβαίας αποδοχής των πιστοποιητικών και σε άλλους τομείς ασφάλειας, εναέριας ασφάλειας, παραδείγματος χάρη άδειες πιλότων ή προσωπικού αέρους, η επίβλεψη της ασφάλειας με ένα γενικότερο τρόπο μέσω ανταλλαγής δεδομένων στα θέματα ασφάλειας. Όσον αφορά τα ατυχήματα, ας πούμε, ή όσον αφορά την επίδοση των ε, αεροπορικών εταιριών. Μένως θέλουμε να καλύψουμε ένα μεγάλο τομέα. Επί της ουσίας τώρα της συμφωνίας, δηλαδή ε, την αμοιβαία αποδοχή των ε, πιστοποιητικών. Η συμφωνία αυτή καλύπτει ένα τεράστιο κενό, διότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία επίσημη, ε, συμφωνία νομικά δεσμευτική, ανάμεσα στην ε, ε, Βραζιλία και σε κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν κάποιες ε, συμφωνίες διοικητικές ανάμεσα σε ορισμένα κράτη-μέλη και την Βραζιλία και είναι πιο, καινούριο αυτό, από το 2004 υπάρχει μια διοικητική ε, συμφωνία, αν θέλετε, μια διοικητική ρύθμιση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εναέριας Ασφάλειας και την, ομόλογο, την υπηρεσία, την ομόλογό της, που είναι υπεύθυνη για την αεροπορική ασφάλεια στην Βραζιλία. Αυτό έχει μια συνέπεια βέβαια. Σημαντική συνέπεια στην αεροναυτική δραστηριότητα, δηλαδή το εμπόριο αεροναυτικών προϊόντων. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να, αναφέρουμε ότι οι εμπορικές ροές ανάμεσα στη, στην ευρωπαϊκή κοινότητα και στη Βραζιλία έχουν αυξηθεί σημαντικά και θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι μέσω των συμφωνιών, των διοικητικών συμφωνιών ανάμεσα στις ε, διάφορες υπηρεσίες ε, μας και την ΑΝΑΚΑ, την αντίστοιχη βραζιλιάνικη δηλαδή, μπορούμε να καλύψουμε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων για τα οποία η παραγωγή πετυχαίνουν σημαντικές οικονομίες, διότι δεν χρειάζεται πλέον μια διπλή πιστοποίηση. Όμως με τη συμφωνία αυτή προχωράμε ακόμα παραπάνω, διότι η συμφωνία αυτή ε, έχει σαν στόχο όλα τα αρμαυτικά προϊόντα να αποτελούν κάποια στιγμή ε, αντικείμενο ε, αμοιβαίας αποδοχής. Ε, επομένως, ε, για, την, για τις αντίστοιχες βιομηχανίες, για τις αντίστοιχες επιχειρήσεις, εταιρείες, ε, το κόστος θα είναι πολύ μικρότερο και θα είναι και λιγότερο δαπανηρές οι υπηρεσίες συντήρησης. Για το σημείο αυτό θα απαντούσα στο ερώτημα που έθεσε η κυρία Λίχτενμπέργκερ, στον τομέα της συντήρησης από την αρχή είπαμε στους Βραζιλιάνους ότι χρειαζόμαστε ε, μια περαιτέρω προσπάθεια από πλευράς τους και η υπηρεσία εναέριας ασφάλειας ε, ήδη μετά, τη συμφωνία, μετά την υπογραφή της συμφωνίας που ε, έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2010 προχώρησε ακόμα παραπάνω η, αποδοχή της έγκρισης, η, όσον αφορά την διαδικασία έγκρισης ε, των ε, εγκεκριμένων, αν θέλετε, ε, συνεργείων θα, λάβει, θα ολοκληρωθεί και θα υπάρξει δηλαδή αμοιβαία αναγνώριση των συνεργείων των συντήρησης στη Βραζιλία μόνο και εφόσον τα στάνταρ φτάσουν ε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, αυτό μπορώ να το διαβεβαιώσω στην κυρία Λίχτενμπέργκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Ευχαριστώ για αυτή την τόσο σαφή απάντηση. Για χρόνια ήμουν υπεύθυνο για τα θέματα εναερίας ασφάλειας ε, στην Ολλανδία και εάν πείτε αν λέτε ότι θα πρέπει να φτάσουν τα στάνταρ τους στα ευρωπαϊκά, νομίζω ότι είναι μια σαφής απάντηση προς την κυρία Λίχτενμπέργκερ. Η κυρία Τικάου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την, όλους τους συναδέλφους ε, και την Κομισιόν βέβαια. Θα ήθελα να σας πω ότι το θέμα της συντήρησης είναι πάρα πολύ σημαντικό επειδή συζητούμε για ένα άνοιγμα της αγοράς στο μέλλον για νέες συμφωνίες πλαίσια και γι' αυτό χρειαζόμαστε πρέπει μάλλον η συντήρηση και αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών να λειτουργεί σωστά η Βραζιλία να μην ξεχνάμε ότι έχει 600 αεροδρόμια παραπάνω από την Ευρώπη καταλαβαίνετε ότι η συντήρηση είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό θέμα Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ όλους. Λέει ο πρόεδρος, ιδιαίτερα τον συνάδελφο Τεξέρα που δεν μίλησε στη γλώσσα του. Ευχαριστώ την κυρία Τικάου ως εισηγήτρια και βεβαίως 9 Φεβρουαρίου είναι η ε, ημερομηνία κατάθεσης των τροπολογιών και από εκεί και πέρα Προχωρούμε. Πάμε στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξη για τον εισηγητή κύριο Ουγγιάς ο οποίο είναι υπεύθυνο για διάφορα για πάνω από ένα θέματα της σημερινή διάταξη, κυρίω για την απαλλαγή του 2009 σε διάφορους οργανισμούς. Έχετε το λόγο κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας μιλήσω για τις, ε, διάφο... απαλλαγές του 2009 για τις διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς. Υπάρχουν κάποια κοινά προβλήματα και θα προσπαθήσω να μιλήσω από κοινού και για τα τέσσερα θέματα που έχουν κοινά σημεία. Ας αρχίσουμε πρώτα απ' όλα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Σκιώδη εισηγητή για την ε, συνεργασία που μου προσέφερε για κάποια ε, θέματα και στα πλαίσια των γνωμοδοτήσεων επί της ουσίας όσον αφορά ε, την ασφάλεια στη θάλασσα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 τα οποία ε, έχουν πρόβλημα εξαιτία τη συμπεριφορά κάποιων υπαλλήλων. Θα ήθελα λοιπόν να ε, διορθωθεί η κατάσταση. Φαντάζομαι ότι οι κανόνες δεν είναι επαρκείς και γι' αυτό θα πρέπει το θέμα αυτό να εξεταστεί σοβαρότερα. Όχι εδώ βέβαια, διότι πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο όλο και περισσότερο μεγενθύνεται. Εάν θέλουμε να υπάρχει εμπιστοσύνη λοιπόν προς τους θεσμούς, θα πρέπει η λειτουργία τους να είναι πιο εύρυθμη. Ε, Σέζαρ. Τώρα θα ήθελα να προσθέσω κάτι για την ε, υπηρεσία Caesar. Είναι μια θετική εκτίμηση σύμφωνα με, την, ε, με το ηλεκτρικό συνέδριο και όλες οι πτυχές είναι κανονικές, νομότυπες κτλ. Πρέπει να σας πω επίσης ότι, έχει, ότι παρά τις δυσκολίες ε, ε, της υπηρεσίας που αυτή τη στιγμή ξεκινάει τη λειτουργία της, ε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ θετικά. Και εφαρμόζεται ο κανονισμός κανονικά από τον Δεκέμβριο του 2008 ο κανονισμός που τροποποιείται την βασική πράξη της κοινή ε, επιχείρησης ΣΕΖΑΡ. Επίσης υπάρχει μια συνεργασία ανάμεσα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και βέβαια υπάρχουν, γι' αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει ε, να αντιμετωπίσουμε θετικά την προσέγγιση της ε, υπηρεσίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τα πάντα είναι τέλεια, υπάρχουν και κάποιες αρνητικές πτυχέ, παραδείγματο χάρη η υπηρεσία αυτή, ο οργανισμό αυτό έχει έναν λογαριασμό 86.800.000 ευρώ, τα οποία συνιστούν παράβαση, παραβίαση της αρχής του ετήσιου χαρακτήρα του προϋπολογισμού. Αυτού του είδους ε, οι επιχει... αυτού του είδους οι, οικονομίες αν θέλετε δεν επιτρέπονται ε, για τους ε, οργανισμούς αυτούς. Δεν ε, έχουν, δεν έχουν λογαριασμούς ταμιευτηρίου οι οργανισμοί αυτοί. Παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποια στοιχεία του ελεκτικού συνεδρίου που αφορούν τους εσωτερικούς ελέγχους που δεν λειτουργήσαν καλά. Όπως επίσης Ζητάμε να υπάρξει ένα σύστημα διαχείρισης έτσι ώστε να ε, καταλογίζονται διάφορες μορφές κόστου σε συγκεκριμένες ενότητες εργασιών και να προσδιορίζονται πηγές χρηματοδότησης για το επιχειρησιακό κόστος. Παρ' όλα αυτά, σε γενικές γραμμές τα πράγματα είναι θετικά, άρα θεωρώ ότι πρέπει να χορηγήσουμε την απαλλαγή. Eh, Ευχαριστώ κύριε Ουτζίας ε, για, την, ε, για τις τόσο λεπτομερείς ε, εξηγήσεις σας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονό ότι έχετε μελετήσει όλου αυτέ τι υπηρεσίε, αυτού του οργανισμού. Πριν δώσω το λόγο στου συναδέλφου, ήθελα να κάνω ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Αναφερθήκατε στην υπηρεσία του σιδηροδρόμων και άκουσα ότι ήταν ανεπαρκής η χρήση. Θέλετε να δώσουμε απαλλαγή για το συγκεκριμένο θέμα ή όχι. Μία αντιευκρίνηση απλώς ήθελα να ζητήσω. Για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων θέλετε να δοθεί απαλλαγή, διότι από ό,τι φαίνεται εκεί είναι η μεγάλη δυσκολία. Μήπως θα μπορούσατε να μπείτε σε προσέγγιση λεπτομέρειες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το συμπέρασμα μου είναι ότι θα πρέπει να χορηγήσουμε την απαλλαγή, διότι το ελεκτικό συνέδριο λέει ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι νόμιμες. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να κάνουμε τους λογιστές. Θα πρέπει να εμείς να κάνουμε μια αξιολόγηση που να ξεπερνάει την ε, λογιστικ, ε, τους λογιστικούς ε, υπολογισμούς. Δεν είμαστε εδώ λογιστές που θα κάνουμε προσθέσεις και αφαιρέσεις. Είμαστε πολιτικοί. Κάνουμε πολιτική αξιολόγηση. Και προφανώς η ύπαρξη δύο εδρών δημιουργεί περαιτέρω κόστος. Εάν όμως από πολιτικής πλευράς ε, επιβάλλεται αυτή η παρουσία των δύο εδρών, ενδεχόμενα θα δώσουμε μια θετική ε, αξιολόγηση. Τώρα, για τα τεχνικά προβλήματα, εμείς θα πρέπει να, και έχουμε υποχρέωση να το εξετάσουμε παραπάνω και να κοινοποιήσουμε και στο Κοινοβούλιο και στην κοινή γνώμη το τι συμβαίνει. Διότι αλλιώς θα ε, είμαστε κι εμείς συνένοχοι για αυτά, για αυτά τα αρνητικά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά συνολικά πιστεύουμε ότι υπάρχουν ε, οι, οι προϋποθέσεις για να χορηγήσουμε την απαλλαγή. Επίσης, μια και μου δώσατε το λόγο, θα πρέπει να αξιολογήσουμε ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνουμε στον οργανισμό για να δούμε την επόμενη χρονιά αν έχουν ξεπεράσει αυτά τα αρνητικά στοιχεία και να ε, μπορέσουμε να είμαστε υπερήφανοι για τη λειτουργία των υπηρεσιών των οργανισμών μας. Δεν ξέρω να πίντησα στο ερώτημά σας, αλλά αν θέλετε μπορώ να πω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα, θα πάρω κι εγώ συνολικά τις, ε, όλες αυτές τις υπηρεσίες. Ε, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή. Πολύ καλή παρουσίαση. Ένα σχόλιο, ένα γενικό σχόλιο. Αυτό το θέμα το οποίο πρέπει να μας, απαλλαγεί, να μας απασχολεί είναι η δημοσιονομική πειθαρχία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι μεταφορές έχουν γίνει. για την, ε, το 65% ποσοστό μεταφέρθηκε, το 65% μεταφέρθηκε στην, ε, το 2010 παραπάνω από το μισό του προϋπολογισμού για την Οργανισμό Αέριας Ασφάλειας για την ασφάλεια των αερομεταφορών. Και μετά έχουμε και κάποια άλλα θέματα αντιμετωπίζονται προβλήματα όσον αφορά την επιλογή του προσωπικού. Ξέρουμε ότι αν τα μέσα μαζικής, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, ε, συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη αυτών των προβλημάτων, νομίζω ότι θα χάσουν την αξιοπιστία τους όλοι αυτοί οι οργανισμοί. Τελευταία παρατήρηση. Σεζάρ. Έχουμε μεταφορά 86 εκατομμυρίων. Πολλά λεφτά. Και δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο. Είμαι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Γι' αυτό τα βλέπω αυτά τα θέματα. Και είναι και πολιτικά τα προβλήματα. Διότι ξέρουμε σε αυτή την οικονομική κατάσταση που επικρατεί. Είναι μεγάλη πολιτική πίεση να περιορίσουμε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και αυτές οι υπηρεσίες που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ούτε το μισό του προϋπολογισμού τους, το 50% του προϋπολογισμού τους, τι θα, τι θα γίνει, δηλαδή το, λογικό είναι να τους πούμε τι χρειαζόσαστε όλο αυτό το προϋπολογισμό όταν δεν χρησιμοποιείτε το μισό. Αλλά τέλος πάντων συμφωνώ με τον ε, εισηγητή ότι θα πρέπει να τις απαλλάξουμε. Γιατί δεν είναι ότι κάνουν λάθος, απλώς, θέλουν απλώς πρέπει να βελτιωθούν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αλκαντράου. Ευχαριστώ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή ε, για τις τόσες λεπτομέρειες που μας έδωσε και ε, κατανοεί απόλυτα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ε, αυτές οι υπηρεσίες, αυτοί οι οργανισμοί. Ε, όντως καταλαβαίνω ότι παρά τα κάποια, τις κάποιες ελλείψεις ε, θα πρέπει να χορηγήσουμε την απαλλαγή. Τώρα όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, όντως εκεί τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα αλλά θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο λόγος, είναι ο λόγος για κάτι τέτοιο. Ίσως θα πρέπει να δώσουμε ε, μεγαλύτερες αρμοδιότητες σε αυτούς τους οργανισμούς, αλλά ίσως να μην τους ε, έχουμε δώσει όλα τα εργαλεία, αν θέλετε, που θα τους επιτρέψουν να ασκήσουν τον καλύτερα τις, ε, τις, τα, τη δουλειά τους. Πρέπει να του δώσουμε τα μέσα, τα, τα αναγκαία μέσα. Ίσως και αυτό άρα να είναι πρόβλημα του Κοινοβουλίου, τη Κομισιόν, του Συμβουλίου. Σε μία επόμενη ανταλλαγή απόψε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων δεν θα πρέπει να μιλήσουμε απλώς και μόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αλλά ίσως θα έπρεπε να δούμε πώς λειτουργεί το όλο σύστημα, συνολικά να το δούμε δηλαδή. Αυτά ευχαριστώ. Ε, Θέλετε να μιλήσετε ε, εξ ονόματος των Πρασίνων. Όχι, να μιλήσει πρώτα κυρία Φώστερ και μετά θα σας το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον εισηγητή για αυτή την τόσο ε, ε, λεπτομερή παρουσίαση που μας έκανε. Ήθελα να πω γενικά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την λειτουργία αυτών των οργανισμών και αυτοί οι οργανισμοί είχαν σαν στόχο να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από, τα, από το υπάρχον καθεστώς, ότι θα, ήταν, ε, ότι θα κοστίζανε λιγότερο, θα ήταν ε, οικονομικά ε, αποτελεσματικοί και θα ήταν, και θα ήταν πιο διάφανοι. Και τι βλέπουμε τώρα όμως, βλέπουμε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο πάντα τουλάχιστον. Και Όντω, όταν πρόκειται για τα πρώτα στάδια τη λειτουργία αυτού του οργανισμού, πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να δεχτούμε ότι δεν θα είναι όλα τέλεια. Για την Ιάσα ήθελα να πω κάτι, ίσως γιατί η Ιάσα, δηλαδή ε, η ασφάλεια των αερομεταφορών ε, και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών είναι πιο ηχηρή αν θέλετε, ακούγεται περισσότερο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η υπηρεσία χρηματοδοτείται από τις εταιρείε κατασκευής αεροσκαφών, από τις αεροπορικές εταιρείε κτλ. Άρα και αυτοί έχουν το λόγο τους, το λόγο, ένα, κάποιο λόγο. Και και για τις διαδικασίες επιλογής των, του προσωπικού. Το ελεκτικό συνέδριο κάνει κάποιες παρατηρήσεις και φαίνεται ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό εκεί. Έχουμε όλο ένα και περισσότερα προβλήματα εκεί. και το πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, ε, Ασφάλειας των Αερομεταφορών ε, έχει αρχίσει να ασχολείται λιγότερο με την ασφάλεια και περισσότερο με τα διάφορα πολιτικά θέματα κτλ. Αυτό είναι ένα μήνυμα όμως το οποίο θα πρέπει να το μεταφέρουμε στην υπηρεσία αυτή ότι θα πρέπει να επανέλθει στο ακαθήκοντά της περισσότερο και να μην ασχολείται με τα να μην, οι, οι, οι εργαζόμενοι εκεί να μην ασχολούνται με διάφορα μικροπολιτικά θέματα. Τώρα για τον Σεζάρ, ο λόγος ύπαρξης του Σεζάρ είναι ε, να είναι πιο αποτελεσματική η να είναι πιο αποτελεσματικές οι εναέρειες κυκλοφορίες στην Ευρώπη. Και θα πρέπει η Επιτροπή Μεταφορών στο Κοινοβούλιο να στείλει ένα σαφές μήνυμα ε, ότι έχετε τα χρήματα στη διάθεσή σας, κάντε τη δουλειά σας. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο θα πρέπει να απευθύνουμε σε όλες τις ε, υπηρεσίες αυτές, σε όλους τους οργανισμούς, ότι πρέπει να κάνουν καλύτερα την δουλειά τους και να μας υποβάλουν καλύτερες εκθέσεις την ε, επόμενη χρονιά. Κυρία Ντυρόν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε δεν μπόρεσα να ακούσω το σύνολο των, ε, των ε, παρατηρήσεων ε, των συναδέλφων, αλλά άκουσα κάποια σχόλια και οφείλω να ομαλογήσω ότι συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που έκαναν οι συνάδελφοι. Για την απαλλαγή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, όντως η απαλλαγή πρέπει να δοθεί και παρά τις, ε, τους μικρούς ενδιασμούς, σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι όντως πρέπει να δοθεί η απαλλαγή. Κύριε Βαντάλε και επευκαιρία τον ευχαριστώ γιατί ε, με αντικατέστησε στην Προεδρία. Πείτε έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ε, ε, στην άδελφο την κυρία Φώστερ πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Εγώ ρώτησα για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων διότι όπως είπα, ελέγχθη. όντως έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος όμως η κατάσταση δεν είναι καθόλου ικανοποιητική, θα έλεγα και διαβάζω την, τις προτάσεις του κυρίου Ούτζιας στο σχέδιο ψηφίσματος. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να είμαστε τόσο ανεκτικοί, αν θέλετε. Και θα υποβάλω τροπολογίες και θα δούμε. Ο κύριος Ρίκη για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Η έδρα είναι στην πόλη που γεννήθηκα, άρα αυτό με ενδιαφέρει παραπάνω. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτη παρατήρηση. Κάποιες ε, σημειώσεις που έκανε ο εισηγητής δείχνουν τη δυσκολία, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο οργανισμός για να ε, λειτουργήσει σε αυτόν τον τομέα των σιδηροδρόμων που είναι δύσκολο, το είδαμε και χτες. Ε, έχουμε 25 χώρες με 25 συστήματα και αυτό έχει δύο συνέπειες. Η πρώτη συνέπεια είναι ότι αυτός ο οργανισμός σιδηροδρόμων καλείται να ε, παρεύει, να αν υπάρχει ένα ατύχημα, ε, κάποιο περιστατικό και τα κράτη-μέλη ζητούν να παρέμβει αυτός ο οργανισμός ε, σιδηροδρόμων. Κάτι το οποίο θεωρητικά δεν θα έπρεπε να κάνει. Ένα πράγμα αυτό. Δεύτερον είναι ότι αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες να προσλάβει προσωπικό. Διότι προσπαθεί να ε, τραβήξει ε, προσωπικό από τις χώρες που, είναι, που έχουν τη μεγαλύτερη εμπειρία στις δρομικές μεταφορές. Αυτές όμως οι χώρες που έχουν μεγάλη εμπειρία δεν αφήνουν το προσωπικό τους να φύγει. Επίσης δεν υπάρχουν ε, δύο έδρες, μία έδρα είναι η στην Βαλονσιέν και στην Λίλε υπάρχει ένα γραφείο. Και η Γαλλία είχε επιχορηγήσει κατά δύο τρίτα την λειτουργία της έδρας, δηλαδή το ενίκιο μειώθηκε κατά δύο τρίτα και με τον τρόπο αυτό αντισταθμίζεται το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το γραφείο υποδοχής στην ΛΙΛ. Άρα για το, το θέμα αυτό δεν ε, πρέπει να δημιουργήσει πρόβλημα και δείτε και την, την αξία, αν θέλετε, ε, στην Βαλονσιάν. Είναι πολύ λιγότερα με το κόστος ε, από οποιαδήποτε άλλη, ε, άλλο οργανισμό. Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις να κάνω. Το ένα είναι η αιτήσιο, ο αιτήσιος προϋπολογισμός των οργανισμών και δεύτερη παρατήρηση για την επιλογή του προσωπικού, διαδικασίες επιλογής του προσωπικού. Αυτό που είπε και ο κύριος Ουτζίας. Όσον αφορά τον ετήσιο προπολογισμό, θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε ανάμεσα στις ε, δεσμεύσεις ε, πιστώσεων και στις δεσμεύσεις πληρωμών. Επομένως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η παρατήρηση του ελεκτικού συνεδρίου αφορά το γεγονός ότι αυτοί οι οργανισμοί κάποιες φορές το 2008-2009 και λόγω της οικονομικής κρίσης μετέφεραν τις πιστώσεις τους στην επόμενη χρονιά. Όλα όμως έχουν γίνει σύμφωνα κανόνες, απόλυτα διάφανοι. Τώρα όσον αφορά ε, για τις διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού. Θα ήθελα να ε, διαβεβαιώσω την Επιτροπή αυτή ότι όσον αφορά την ένσα, η έλλειψη... Το πρόβλημα ήταν η έλλειψη εσωτερικού ε, εκπροσώπων του, της Επιτροπής Προσωπικού κατά τις διαδικασίες πρόληψης. Ε, δεν υπήρχε τότε Επιτροπή Προσωπικού και ε, νομίζω ότι τώρα που δημιουργήθηκε λύθηκαν το πρόβλημα. Άρα ε, υπάρχει τώρα η παρουσία για κάθε πρόσληψη εκπροσώπων της Επιτροπής Προσωπικού. Το πρόβλημα είναι να βρούμε τα άτομα τα οποία είναι κατάλληλα να κάνουν την επιλογή. Αυτό είναι τη μεγαλύτερη, αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει η υπηρεσία. Το πρόβλημα είναι ότι είναι ε, οι εμπειρογνώμονες, ιδίως για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, είναι εκεί μέχρι, ε, για, λίγα, λίγα χρόνια και μετά φεύγουν. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί κόσμος να πάει στη Βαλονσιέν, γιατί η Βαλονσιέν μιλάμε, όχι για τη Λίλου. Ευχαριστώ κύριε Μπονούτσι. Ο Δήμαρχος της Βαλονσιέν, είμαι σίγουρος ότι θεωρεί ότι είναι εξαιρετικό το, εξαιρετική πόλη Λοιπόν, για, την έκθεση UGS, ε, τροπολογίες μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, 28 Φεβρουαρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή Μεταφορών, 28 Μαρτίου από την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών και μετά θα περάσει στην ε, Ολομέλεια. Για μας η προθεσμία υποβολής τροπολογιών 1η Φεβρουαρίου. Επόμενο σημείο αφορά την ε, απαλλαγή της ε, Κομισιόν. Κύριος Γκρός. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι πρόκειται εδώ για την απαλλαγή, για το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Θα ήθελα όμως, θα ήθελα πριν μπω σε λεπτομέρειες να πω κάτι που ακούστηκε και προηγούμενα. Η... Αν δεν έχει τηρηθεί ο ετήσιος δεν ε, μπορεί κανείς να... Ε, ε είναι ε, να τιμωρήσει αν θέλετε γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να πρόκειται για λάθος αλλά ε, αν αυτοματοποιήσουμε ορισμένα πράγματα θα δημιουργήσουμε περισσότερα προβλήματα από ό,τι θα λύσουμε εφόσον διατηρείται η διαφάνεια δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τώρα από εκεί και πέρα να πω ότι για τα διευρωπαϊκά δίκτυα είχαμε 934 εκατομμύρια υποχρώσεις 930 περίπου χιλιάδες ε, πληρωμές ε, χρήση των κονδυλίων 100% ε, ε, στην έκθεση επίσης αναφέρονται οι διάφοροι οργανισμοί τους οποίους δεν θα αναφέρω ξεχωριστά και όσον αφορά τα θετικά μηνύματα αναφέρεται και ο Γκαλιλαίο που έχει ψηλό ποσοστό πρόφιλ χρήσης αλλά όπου κάπου λέγεται ότι η αποτελεσματικότητα του προγράμματος δεν μπορεί να μετρηθεί μέσω της χρησιμοποίησης των κονδυλίων. Πρέπει να περάσουν μερικά χρόνια. Ε, λίγο. Τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι την Κομισιόν. Για τον Μάρκο Πόλο, από ό,τι θυμάμαι, η τα κονδύλια του Μάρκο Πόλο τα ενέκρινε και η Επιτροπή Μεταφορών εδώ. Ήταν μια καλή πρωτοβουλία θεωρήσαμε. Αλλά μετά τα ποσοστά απορρόφησης και χρήσης ήταν πολύ μικρά και γι' αυτό αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε μήπως τα κριτήρια δεν ήταν σωστά. Τώρα εδώ διαβάζω στην έκθεση και θα ήθελα να μου εξηγήσει η Κομισιόν ότι έχουμε αυξημένη απορροφητικότητα στα κονδύλια του Αμάρκο Πόλο αλλά ε, ότι χρησιμοποιήθηκαν μόνο 50% των κονδυλίων. Δηλαδή τι έγινε, κονδύλια του Μάρκο Πόλο διατέθηκαν για άλλο σκοπό. Και κάτι τι άλλο, στην Επιτροπή λέμε πολύ συχνά ότι η, για τα ευρωπαϊκά δίκτυα ιδιαίτερα ε, ε, ότι και η χρήση η απορροφητικότητα εκείνων των κονδυλίων και για άλλα θέματα αυτά πάνε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης η αυτή είναι η πιο αρμόδια κτλ. Ε, εδώ μπαίνουν τα διευθυντικά ταμεία στο παιχνίδι και ε, κάπου ε, η μπερδεύονται τα πράγματα. Εκείνο το οποίο για μένα είναι κακό είναι ότι ορίζουν, προτιμώνται προγράμματα και χρηματοδοτούνται προγράμματα ε, ακόμη και αν η χρηματοπιστωτική ανάλυση που γίνεται στην αρχή είναι κακή. Και δεν δε γίνεται σωστά η ανάλυση. Θα έλεγα λοιπόν ότι η Επιτροπή ε, προπολογισμών και ελέγχου των προπολογισμών εδώ στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να ε, παρακολουθεί λίγο παραπάνω τα, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης γιατί εδώ υπάρχουν ε, κάποια δεν λέω ότι συμβαίνουν σκανδαλώδη πράγματα αλλά ε, δεν είναι πολύ καλή Τώρα κάτι τι άλλο ε, γιατί διάβασα και την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και ε, ε, των συντονιστών α, μάλλον το ελεκτικό συνέδριο στην δική έκθεση δηλαδή, διαπιστώνει ότι οι συντονιστές είχαν πολύτιμη συμβολή ε, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Νομίζω πρέπει να το χαιρετήσουμε. Από εκεί και πέρα όμως αναφέρεται ότι για έργα προτεραιότητας στις ε, μεταφορές και στην, ε, στις υποδομές ε, μπορούν κάποια πράγματα να βελτιωθούν. Πέρα από τα παράπονά μου αυτά και πέρα από την απάντηση που θέλω να μου δώσει για τον Μάρκο Πόλο Κομισιόν υποστηρίζω να δοθεί απαλλαγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Ο κύριο Αλκαντράουι, όχι. Η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η κυρία Γιάντσεν που είναι σκιώδη συγγήτρια δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα και γι' αυτό μου ζήτησε να πάρω εγώ το λόγο. Οι γενικές θέσει θέσεις της ε, συμπίπτουν με αυτές του κυρίου Γκρεός τα αναφέρει και εκείνη ότι το Μάρκο Πόλο πρέπει να μελετηθεί υπεραιτέρω να παρακολουθηθεί καλύτερα και όπως είπε και ο κύριος Γκρεός λέει ότι είναι μεγάλη η ανάγκη για καλύτερο συντονισμό μεταξύ της πολιτικής μεταφορών και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το αναφέρει και αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια η αρμόδιοι επίτροποι είναι σε επαφή υποθέτω αλλά καλά κάνει το Κοινοβούλιο και ζητάει, τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερο συντονισμός. Η κυρία Γιάννησεν μπορεί να έχει και άλλες παρατηρήσεις να κάνει, ίσως θα είχε αν ήταν εδώ, αλλά σε γενικές γραμμές συμφωνεί με τον κύριο Γκρόρς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντουιρό. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ και στον τον κύριο Γκρός για την έκθεσή του. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που έγινα. Τώρα ειδικά για τον Μάρκο Πόλο να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτη για την πράγματι για το συντονισμό μεταξύ του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Συνοχής και τα λοιπά ε, χρειάζεται καλύτερο συντονισμός αλλά νομίζω ότι είστε και θέμα ενημέρωσης και διαφάνειας δεν είναι μόνο θέμα συντονισμού ε. Ε, ε, είπατε ότι πολλές φορές δεν ε, υπάρχουν όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες αλλά εγώ νομίζω ότι τα, η διαφάνεια και ε, είναι σημαντικό που θα πρέπει να το σημειώσουμε. Δεύτερη παρατήρηση που απευθύνω προς την Κομισιόν. Η Κομισιόν θα ήθελα να ξέρω τι λογαριάζει να κάνει με τις παρατηρήσεις που κάναμε που, έγιναν για τα έγιναν κάποιες παρατηρήσεις κάναμε κάποιες παρατηρήσεις για κάποια κονδύλια για τις μεταφορές η Κομισιόν τι κάνει με αυτές τις παρατηρήσεις ε? δεν λέω ότι επηρεάζεται η απαλλαγή αλλά τις έχει τις παρατηρήσεις μετά η Κομισιόν τι λογαριάζει να κάνει δηλαδή να τις λάβει υπόψη ε, να κάνει κάποια πράγματα λόγω αυτών των παρατηρήσεων κτλ. Ο κύριος Μπράτμπορ Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ το Ματιό Γκρός για τη δουλειά που έκανε και να πω ότι συμφωνώ με πάρα πολλά από τα σχόλια που έγιναν. Όμως πρόεδρε Είμαι, βρίσκομαι στη θέση που βρίσκομαι εδώ και 200 και εδώ και 12 με συγχωρείτε χρόνια. Κάθε φορά παίρνουμε μια έκθεση, κάνουμε τις επικρίσεις μας, λέμε ότι ε, πολλά πράγματα θα πρέπει να βελτιωθούν, αλλά λέμε ε δεν πειράζει μωρέ δώσ' τους την απαλλαγή. Ε, Οφείλω λοιπόν να πω πρόεδρε χωρίς να είμαι άδικος στο, για το για την Επιτροπή Μεταφορών δεν είναι χειρότερη σε αυτό αλλά οφείλω να πω όμως όπως είπε και ο κύριος Γκρός δικαίως ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει επιγόντως να μελετηθούν παραδείγματο χάρη περιθώρια σφάλματος ε. ε, πρέπει να βελτιωθούν τα πράγματα αν δούμε εδώ η Κομισιόν μιλάει για ένα προϋπολογισμό δύο δις Δύο δις ε, λιρών παραδείγματος χάνει και ακόμη και αν το περιθώριο σφάλματος είναι μόνο 5% όπως λέγεται εδώ αυτό είναι 100 εκατομμύρια λίρες του φορολογούμενου που πρέπει κάπου να δικαιολογηθεί δεν είναι λοιπόν τόσο απλά τα πράγματα και που δεν είναι λόγο υπονοώ ότι ε, εδώ ε, ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος που έχει συμβεί ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά κάνω μια γενική παρατήρηση έχουμε δημοσιονομική πειθαρχία έχουμε δημοσιονομική λογοδοσία και το λέμε, μιλάμε για ένα σφάλμα 100 εκατομμυρίων λιρών τώρα το άλλο που είπε ο κύριος Γκρός για τις διαδικασίες επιλογής όντως πρέπει να γίνεται η επιλογή με πολύ με διαφορετικό τρόπο και με πολύ πιο στέρεο οικονομικό σχεδιασμό διότι εδώ αν δεν κάνω λάθος απλώς μοιράζονται έτσι ελαφρά την καρδία τα κονδύλια χωρίς κανείς να μελετά το πώς θα χρησιμοποιηθούν τελικά και κάτι τι άλλο που σχετίζεται με το προηγούμενο, αλλά που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Τις μελέτες σκοπιμότητας. Ξοδεύουμε χρήματα για σχέδια και προγράμματα ε, τα οποία δεν θα αποφέρουν μεγάλο όφελος. Γιατί πρέπει να ε, εφαρμόσουμε κάποιους κανόνες χρηστής διαχείρισης, να κάνουμε κάποιες μελέτες, ε, κόστους οφέλους και μετά να προχωρούμε πιο σοβαρά. Ο κύριος Μενούτσι. Ε, Ευχαριστώ. Να απαντήσω πρώτα πρώτα για το Μάρκο Πόλο. Γιατί έτσι το ερώτημα. Το πρόγραμμα Μάρκο Πόλο συνδέεται στενά με την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών και θαλάσσιων μεταφορών. Τα κονδύλια καταβάλλονται σε, ανάλογα με τη μετακίνηση τόνου το, κάποιου βάρους, κάποιων τόνων ανά απόσταση, ανά χιλιόμετρα και το 2008, το 2009 αυξήθηκε η απορρόφηση των κονδυλίων του Μάρκο Πόλο. Ε, ε, ζητή, έγιναν αλλαγές και ζητήθηκε να καταργηθεί και η ε, προκαταβολή η οποία δινόταν παλιά. Αντιμετωπίσαμε την ε, πολύ δύσκολη κατάσταση να έχουν δεσμευθεί κονδύλια για να δοθούν και να μην μπορούν να γίνουν πληρωμές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τέλος πάντων, έκτοτε έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, φέτο είναι καλύτερα. Ε, τα ποσοστά εκτέλεση έχουν αυξηθεί. Λάβετε υπόψη σας βέβαια ότι έγινε αναθεώρηση του κανονισμού το 2009 και έτσι ο μηχανισμός έγινε πιο κατανοητός, πιο ελκυστικό από οικονομική απόψεω. Για το 2011 περιμένουμε να επανέλθουμε σε πολύ, καλή, σε πολύ καλά επίπεδα. Τώρα για τα διευρωπαϊκά δίκτακα, δίκτυα, γιατί έτσι και σχετικές ε, ερωτήσεις και για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Λάβετε, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Ε, λάβετε υπόψη σας ότι τα, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά κύριο λόγο διοικείται από το, την τοπική αυτοδιοίκηση, ε από τις τοπικές κυβερνήσεις τα κράτη-μέλη και ε, Βεβαίω και από εκεί και πέρα εφαρμόζονται και πληρώνονται τα σχέδια ένα προς ένα. Έχουμε προγραμματισμό βέβαια πολυετή, έχουμε και αιτήσιο. από εκεί και πέρα όμως ε, έχουμε και κατηγορίες σχεδίων ε, υψηλής προτεραιότητας, μέσης προτεραιότητας και χαμηλής προτεραιότητας. Τώρα όσον αφορά το περιθώριο σφάλματος, είναι αλήθεια, είναι μεταξύ 2 και 5%, λίγο λιγότερο από 5%. Φέτος είμαστε λίγο πάνω στο από το 2,4-2,6%. Τι γίνεται τώρα, πώς το υπολογίζουμε αυτά, τι κάνουμε. Κάνουμε τους ελέγχους, τους ενδιάμεσους και τους εξπόστ. Ε, ενημερώνουμε, κάνουμε ε, ad hoc επισκέψεις, κάνουμε προληπτικούς ελέγχους. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε στους δικαιούχους ποιοι είναι οι κανόνες, ε, πώς πρέπει να εφαρμόζονται και σε τελευταία ανάλυση πριν να υποβληθεί οποιοδήποτε δήλωση κόστους προσπαθούμε να βοηθήσουμε το δικαιούχο, δικαιούχο να καταλάβει τα πράγματα και να καταλάβει τι ακριβώς μπορεί να αξιώσει, μπορεί να ζητήσει. Έτσι τα λάθη μειώνονται και άρα και το συνολικό περιθώριο σφάλματος ελπίζουμε να μειωθεί στο μέλλον. Καταβάλουμε πάσα προσπάθεια, αλλά δεν θέλουμε να τιμωρούμε, ε, να κυνηγούμε τους δικαιούχους after, ε, ανεφλόγου. Θέλουμε να καταλάβουν και αυτοί για να μπορούν να μην κάνουν λάθη στο μέλλον. Ωραία κύριος Κρός. Με δύο λόγια, κοιτάξτε να δείτε. Η κυρία Ντουράου μίλησε για τη διαφάνεια. Ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα να βάλω εδώ κάτι για την διαφάνεια. Κανένα πρόβλημα δεχτώ την πρότασή τώρα για τα λάθη και τα περιθώρια ασφάλματο και τα ε, καλό θα ήταν να συνεχίσουμε να διατηρήσουμε την ε, ε, παρατήρηση που έχουμε κάνει εδώ γιατί μας λέει η Επιτροπή ότι στο μέλλον θα βελτιωθούν τα πράγματα αλλά δεν πειράζει ίσως καλύτερο θα ήταν να διαγράψουμε του χρόνου και για την ενημέρωση όπως και η κυρία Τουρό. εμείς σαν κοινοβούλιο πρέπει να ενημερωνόμαστε άμα βλέπουμε ότι έγιναν δαπάνες που δεν έπρεπε να γίνουν και ότι ε, ζητείται επιστροφή των αχρεώσεων εφαρμοστεί τους ποσών. Δεν λέμε ότι αυτό είναι απάτη, είναι σκάνδαλο, αλλά θα πρέπει να ενημερώνονται οι πάντες γι' αυτό, να υπάρχει καλύτερος συντονισμός, να υπάρχει καλύτερη διαφάνεια. Τώρα αν η απόφαση θα έρθει από πάνω ή από κάτω δεν ξέρω, αλλά οι, δια, οι επενδύσεις ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών και των διευρωπαϊκών δικτύων θα πρέπει να γίνονται με ε, πιο στέρεα κριτήρια. Ε, λοιπόν αυτά όλα πρέπει να είναι απαιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διατηρούμε ακόμη την παρατήρηση και ίσω διαγράψουμε του χρόνου αν βελτιωθούν τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. 1η Φεβρουαρίου ναι, η, ε, η ημερομηνία κατάθεσης των τροπολογιών 28 Φεβρουαρίου ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή και βλέπουμε από εκεί και πέρα για την Ολομέλεια. Λοιπόν, 1η Φεβρουαρίου ημερομηνία κατάθεσης των τροπολογιών. Α, ξέχασε τον κύριο Ουγγίας. Έπρεπε να του είχα δώσει το λόγο. Ε, να δούμε αν θέλει να πάει κάτι τι, μετά από την Κομισιόν. Έχετε το λόγο. Όχι, εντάξει, δεν χρειαζόταν. Απλώς κατά την απουσία σας συζητήσαμε όλα τα θέματα ε, και τις λεπτομέρειες. Συμφωνώ βέβαια για, ε, για τα, όσα τα όσα είπατε. Θα περιμένουμε τις τροπολογίες και θα δούμε. Κάτι άλλο δεν θέλω να πω. Ούτζα είμαι είναι το όνομά μου στα Ιταλικά, έτσι, Ούτζα. όχι Ούγγιας. Το καταλαβαίνω ότι για του ε, Βρετανού και για τους Γερμανούς ενδεχόμενα είναι δύσκολο. Αλλά εδώ η φίλη μου η Γερμανίδα τα καταλαβαίνει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Θα προσπαθήσω να το λέω σωστά το όνομά σα στο μέλλον. Πολύ ωραία. Άλλα θέματα που θέλετε να συζητήσουμε. Εάν όχι, να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 14 Φεβρουαρίου του Αγίου Βαλεντίνου. Και μετά θα έχουμε και τη συνάντηση στο, στο Στρασβούργο με τον Επίτροπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προσπάθειές σας. Πέρασε συνεδρίαση να ε, υπενθυμίσω στους συντονιστές ότι θα πρέπει να είναι εδώ στις 12. Ευχαριστώ.